Αύριο θα γίνει ψηφοφορία επί της έκθεσης αυτής και περνάμε τώρα στην μία σύντομη παρουσία της έκθεσης Άννα Ζαμπόλσκα για την ομαλυψία με βάση το φύλλο και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη συνεργασία τους, για την ε, έκθεση αυτή ε, πρωτοβουλίας. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών ήταν το αποτέλεσμα μιας ευρύτατη συζήτηση που έγινε. Ε, και οι άντρες και οι γυναίκες που ε, πλέκονται ε, στο θέμα, με το θέμα της αλληλεγγύης μεταξύ των ε, γενεών αξίζουν υποστήριξη διότι συμβάλλουν στη δημιουργία πλούτου και στο γενικότερο καλό. Δυστυχώς η εργασία αυτή δεν περιλαμβάνεται στις εθνικές στατιστικές και στα λογιστικά βιβλία και γι' αυτό αυτοί οι άνθρωποι, οι άντρες και οι γυναίκες είναι αντικείμενο διακριτικής μεταχείρισης. Όλοι οι άντρες και γυναίκες, όλοι όλοι οι άνθρωποι θα έπρεπε να είναι ε, σε θέση να επιλέγουν τον ε, τρόπο εργασίας τους και η κοινωνία θα πρέπει να τους ε, ανταμείβει γι' αυτό και να μην ασκεί διακριτική μεταχείριση εις βάρος τους γιατί απλώς δεν πρόκειται για εργασία στην αγορά. Αυτό είναι θέμα και ισότητας των φίλων και αλληλεγγύης μεταξύ των γενναιών. Το θέμα της έκθεσής μου ε, αφορά την ε, απασχόληση ε, στην Ευρώπη του μέλλοντος. Ίσως η συζήτηση αυτή είναι πολύ τεχνική, αλλά έχει και μια ανθρώπινη διάσταση. Ο καθένας από εμά μπορεί να βρει τον εαυτό του μέσα σε αυτή την έκθεση, γιατί όλοι έχουμε οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις. Το να προσπαθήσει κανείς να ερμηνεύσει τον όρο αλληλεγγύη μεταξύ ε, των γενναίων και φροντίδα των παιδιών είναι ε, ε, μια μεγάλη προσπάθεια. Γι' αυτό μπορεί να καλύπτει και την φροντίδα των ηλικιωμένων γονέων και άλλων μελών της οικογένειας. Επίσης, αλληλεγγύη σημαίνει και εκπαίδευση των παιδιών να σέβονται τη ζωή, το περιβάλλον θέμα βασικά κοινωνικής δικαιοσύνης και είναι η βάση για το μέλλον της Ευρώπης και για το κοινό καλό όλων των πολιτών. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί αυτός ο πλούτος με πολύ συγκεκριμένο και ρητό τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ε, εξασφαλίσει το ε, πολιτικό πλαίσιο για να επιτεθεί αυτός ο στόχος. Οι γυναίκες ε, συνήθως είναι οι πρώτες που ε, εμπλέκονται σε θέματα αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και γι' αυτό ε, τις γυναίκες αφορά κατά κύριο λόγο ε, η έκθεση αυτή. Οι οικονομολόγοι χρησιμοποιούν μαθηματικά μοντέλα που αποδεικνύουν ήδη την αξία της κατοίκων εργασίας και δημογραφικές και οικονομικές μελέτες δείχνουν ότι η συμβολή των γυναικών είναι πολύ σημαντική στο ΑΕΠ. Αυτά βέβαια τα δεδομένα αφορούν το παρελθόν. Πρέπει να κοιτάξουμε προς το μέλλον για να δημιουργήσουμε ε, τις κατάλληλες συνθήκες για αυτούς τους ανθρώπους που ε, εργάζονται στο επίπεδο της αλληλεγγύης μεταξύ των γενναιών. Και Πρέπει να το κάνουμε αν εννοούμε σοβαρά την πολιτική της μη διακριτικής μεταχείρισης. Το κόμμα μου ε, με υπερηφάνεια υποστηρίζει τις αρχές της μη ε, διακριτικής μεταχείρισης, της ισότητας των φύλων και της συμπληρωματικότητας ε, του ρόλου ανδρών και γυναικών. Αγαπητοί συνάδελφοι, η έκθεση αυτή είναι το αποτέλεσμα της διαβουλή με πολλές γυναίκες, με πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Επίσης έχω σεβαστεί ε, τις ε, ε, θέσεις των τριών μεικτών ομάδων, διακομματικών ομάδων στην, στο Κοινοβούλιο. Έχει εγκριθεί ομόφωνα από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών η έκθεση αυτή και ζητώ την υποστήριξή σας. Πρόεδρε, νομίζω ότι η κυρία Ζαμπόσκα επιτέλεσε πάρα πολύ έργο γιατί το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλης σημασία στην κοινωνία μας. Αυτή η εξάρτηση αποκτά λένε για περισσότερη σημασία λόγω του δημογραφικού προβλήματος της γύρνησης του πληθυσμού και γιατί και τους ανήλικους και τους ε, υπέργυρους γυναίκες τους περιποιούνται επομένως θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα που να βοηθήσουν τις γυναίκες που να μπορέσουν να μείνουν κοντά στην αγορά εργασία, να βελτιωθούν επίση και οι συνδίκε οικογενειακού βίου και να υπάρχει καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και οικογενειακού βίου. Τώρα, όσον αφορά το τι ισχύει όσον αφορά τα εξαρτώμενα μέλη, ήδη έχουμε προτείνει δράσεις. η άδεια ε, πέρασε από τη διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά την, το συμβασμό επαγγελματικού και ε, οικογενικού βίου. Επίσης είπαμε ότι θα πρέπει να βοηθούν οι υπέργυροι να μην γίνεται κακό μεταχείριση και είπαμε ότι είναι δυνατόν να ληφθούν κάποια μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και να επιταχύνουμε τις εξελίξεις για εξυγχρονισμό των υποδομών και των υπηρεσιών. νέα πολιτική συνοχή μέσω του Κοινωνικού Ταμείου και πρωτοβουλίες συγχρηματοδότησης και σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο. Ανοιχτή μέθοδος συντονισμού για κοινωνική πρόνοια και κοινωνική ένταξη και να προσέξουμε ιδιαίτερα τις συντάξεις των ισχυρισμών τους, να λεφθούν υπόψη νέες μορφές εργασία να καλυφθούν τα εξαρτώμενα μέλη Οπότε, όπως λέτε, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, ε, ασχολούμεθα με το θέμα και περιμένουμε πώς και πώς την περαιτέρω συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Το οποίο και συγχαίρουμε για αυτό το σημαντικό έργο. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Αύριο τρίτη θα γίνει η ψηφορία. Και τώρα. Α, όμως, η κυρία Παγιωτοπούλη Κασιώτου έχει δει το λόγο. Πρόεδρε. Ε, ήθελα να παρατηρήσω ότι σε αυτή την έκθεση που ψηφίστηκε ε, με ε, απόλυτη πλειοψηφία στην ε, επιτροπή γυναικών υπάρχει ένα ψήφισμα ε, εναλλακτικό που έχει κατατεθεί από κάποιους συναδέλφους και θα κληθούμε να ψηφίσουμε αύριο ανάμεσα στο ψήφισμα των συναδέλφων και στο ψήφισμα που έχει εγκριθεί από μια επιτροπή του κοινοβουλίου. το ένα καταρρύπτει το άλλο. δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό το εναλλακτικό ψήφισμα στην ολομέλεια. δεν μπορούμε ούτε να ακούσουμε τους συναδέλφους που το έχουν έχουν καταθέσει ούτε εμείς να εκφραστούμε γι' αυτό. Ε, είναι μια ατέλεια του νέου κανονισμού που πρέπει να λάβετε υπόψη. ευχαριστώ. Euh, ναι, ισχύει αυτό που είπα και πριν για την κυρία Ντόιλ. Επικαλούμεθα το άρθρο 45 και επομένω το πλαίσιο είναι αυστηρό όσον αφορά το χρόνο αγόρευση. Διότι δεν τον Πρόεδρο να απεφάσισε έτσι να αντικυπηρεθεί αυτό το θέμα. μια αυτού του άρθρου. Φυσικά και θα πρέπει ο κανονισμό να γίνει τέτοιο τόσο ώστε να επιτρέπει περισσότερη ευελιξία. Δεν μπορούμε τώρα όμω να αλλάξουμε τον κανονισμό και θα λάβουμε απλώ υπόψη την παρατηρήση σα τελευταίο τώρα. Σημείο τη σημερινή διάταξη είναι σύντομη εισήγηση εκθέσεω Harbor. Προεμπορικέ δημόσιε συμβάσει, πρόθεση και ονοτομή στην εξασφάλιση βιώσιμων και ποιοτικών δημοσίων υπηρεσιών στην Ευρώπη. Έχει το λόγο, κύριε Χάρμπορ. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευτυχώ που έχουμε εδώ την κυρία Ρέντινγκ από την Κομισιόν απόψε